Η ημέρηση διάταξη προβλέπει την ψηφοφορία της έκθεσης του κυρίου Κράσιλ Ντέρφελ για τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Ο κύριος Κράσιλ Ντέρφλερ θα υποβάλει τρεις προφορικές τροπολογίες. Έχετε το λόγο κύριε Σιγητά. Θα εξετάσουμε ξεχωριστά κάθε ε, μία προφορική τροπολογία. Κύριε Ισηγητά, παρουσιάστε μας παρακαλώ την πρώτη προφορική τροπολογία. Κύριε Πρόεδρε, λόγω των ε, διεθνών γεγονότων πρέπει να κάνουμε δύο τεχνικές ε, διορθώσεις. Το εκτιμώντας L, το όνομα του Μουαμάρ Αλκαντάφη θα πρέπει να αφαιρεθεί γιατί βεβαίως ε, και στο άρθρο 24 το ίδιο. Ο δε Σαΐφ Αλισλάμ Καντάφη ο ιός του και ο Σανίφα Λασλούμι της ε, Λιβύης επίσης δεν είναι στι που είχαν και παρακάτω θα πρέπει να συμπληρωθεί στο διεθνές, ε, σύμφωνα με το διεθνές ε, ανθρωπιστικό δίκαιο και στη διεθνή δικαιοσύνη. Νομίζω δε πως ερχόμαστε την κατάλληλη στιγμή με αυτή την έκθεση. Αν δούμε την κατάσταση στην Συρία πρέπει να πούμε πως όλοι αυτοί οι δολοφόνοι και τύρανοι θα πρέπει να νιώθουν πως υπάρχει μία δαμόκλειο σπάθη η οποία επικρέμεται πάνω τους και πάντα υπάρχει η δυνατότητα να αποδοθεί δικαιοσύνη. Ευχαριστώ δε όλους τους συναδέλφους και τους συντονιστές για τη στήριξή τους. Σας ευχαριστούμε κύριε εισηγητά. Ο εισηγητής παρουσίασε ταυτόχρονα και τις τρεις προφορικές τροπολογίες. Υπάρχουν αντιρρήσεις. Θέλει κανείς να αντιταχθεί, α σηκωθεί παρακαλώ από τη θέση του. Α σηκωθεί όρθιος, δεν βλέπω κανέναν. Οπότε υπάρχει συμφωνία για να ψηφίσουμε τις τρεις προφορικές τροπολογίες. Ψηφίζουμε ονομαστικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνονται. Συγχαρητήρια, συνάδελφε. Η επόμενη ψηφοφορία αφορά την έκθεση του κυρίου Κουμουτσάκου για την περαιτέρω ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής. Το σχέδιο κανονισμού πρώτα. Πρώτο μπλοκ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα καταπίπτει. Ψηφίζουμε την ούτως που τροποποιηθεί στα πρόταση επιτροπής. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συγχαρητήρια κύριε Σιγητά. Ψηφίζουμε το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Ψήνεται. Εγκρίνεται. Ευχαριστώ τον εισηγητή. Επόμενο θέμα, έκθεση Ψεζίνα για το πρόγραμμα και πλαίσιο δραστηριοτήτων πυρηνικής έρευνας και εκπαίδευσης Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας. Ε, εξετάζουμε το ψήφισμα, το σχέδιο ψηφίσματος. Ε, 22 επι, ε, τροπολογίες Επιτροπής ε, Ενέργειας υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 3 με ονομαστική ψηφοφορία, άρχιτη ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνονται. Τροπολογία 8, ονομαστική ψηφοφορία, άρχιτη ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι τέλο ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 34. Ψηφοφορία κατά τμήματα με ονομαστική κλίση. Δύο τμήματα ονομαστικά. Άρχεται η ψηφοφορία για το πρώτο τμήμα. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται το πρώτο τμήμα. Δεύτερο τμήμα, ονομαστικά έρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Απορρίπτεται. Τροπολογία 14. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 30. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 30. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 16. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 35 ονομαστική ψηφοφορία, άρχιτη ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 21. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 36, ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 31, ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 32. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχιτη ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 33 με ονομαστική κλίση. Άρχιτη ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε την ούτως τροποποιηθής απρόταση επιτροπής. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια κύριε Ψιζίνα και σας ευχαριστούμε. Επόμενη ψηφοφορία αφορά τις προτάσεις ψηφίσματος με θέμα τη συνάντηση κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών που θα λάβει χώρα στις 28 Νοεμβρίου του 2011. Κοινό ψήφισμα πέντε πολιτικών ομάδων. Τροπολογία 1. Ο κύριος Μπρόκ ζήτησε το λόγο, παρακαλώ. Κύριε Μπρόκ. Κύριε Πρόεδρε, εδώ πέρα έχω κάνει ένα λάθος. Θα ήθελα να συστήσω ε, στην ομάδα μου να υπερψηφίσει την τροπολογία 1. Καλώς. Ας ψηφίσουμε. Τροπολογία 1. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 8. Ψηφοφορία κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 11. Ψηφοφορία κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 2. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 14. Ψηφοφορία κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα. Ποιο είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 22. Η κυρία Λούτφορτ ε, έχει προφορική τροπολογία για την παράγραφο 22. Έχετε το λόγο κυρία Λάτφορτ. Κύριε Πρόεδρε. Πρόκειται για τροπολογία η οποία πραγματικά αντιπροσωπεύει την αλήθεια, τα γεγονότα. Γιατί λαμβάνει υπόψη τη ε, τη δήλωση της Επιτροπής ε, σχετικά ε, με την ολοκλήρωση της συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με το PNR σε συνέχεια της διαδικασίας της 5 Μαΐου του 2010. Η αυθεντική διατύπωση τελικά ήταν πλέον πεπαλαιωμένη γιατί έχει προχωρήσει η Κομισιόν σε ανακοίνωση και επομένως στην ουσία απλώς αντιπροσωπεύει ε, την πραγματικότητα. Δεν έχει καμία υποκειμενικότητα. Ευχαριστώ. Έχει κανείς αντίρρηση για την προφορική τροπολογία? Δεν βλέπω αντιρρήσεις. Ψηφίζουμε την παράγραφο 22. Ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές, κατά συγγνώμη, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 4. Ποιος είναι υπέρ. Συγγνώμη, υπάρχει μια πρόταση για ηλεκτρονικό έλεγχο. Όχι, όχι, εντάξει, εντάξει. Τροπολογία 4. Τότε ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 4. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Μετά το 25, ο κύριος Μπροκ θα υποβάλει προφορική τροπολογία για το 25α. Έχετε το λόγο κύριε Μπροκ. Κύριε Πρόεδρε, οι συνάδελφοι σε διάφορες επιτροπές ε, προετοιμαζόμενοι για την ε, Σύνοδο Κορυφής με Τσίπα έχουν υποβάλει πάρα πολλές χρήσιμες ε, τροπολογίες οι οποίες βεβαίως δεν μπορούν να γίνουν όλες δεκτές αλλά με την άδειά σας θα ήθελα να ενσωματωθούν αυτές σε μία προφορική τροπολογία λαμβάνει υπόψη τις συγκεκριμένες προτάσεις των διαφόρων επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ζητά από την Ευρωπαϊκή ε, από την αντιπροσωπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να χρησιμοποιήσει αυτές. Έχει κανείς αντιρρήσεις για την προφορική τροπολογία? Δεν βλέπω ενστάσεις. Μάλλον χαρά και επιδοκιμασία διαπιστώνω. Ψηφίζουμε μετά το 25, το 25α. Ποιος είναι υπέρ? κατά αποχές εγκρίνεται με την προφορική τροπολογία. Ψηφίζουμε τώρα το κοινό σχέδιο ψηφίσματος. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και ευχαριστώ τους συναδέλφους γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό το κοινό ψηφίσμα. Επόμενη ψηφοφορία προτάσεις ε, για το ανοιχτό διαδίκτυο και ουδετερότητα του διαδικτύου στην Ευρώπη. Ψηφίζουμε το σχέδιο ψηφίσματος γιατί δεν έχουν κατατεθεί τροπολογίες. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Επόμενο θέμα. Προτάσεις ψηφίσματος για την απαγόρευση των πυρομαχικών διασποράς. Κοινό σχέδιο ψηφίσματος πέντε πολιτικών ομάδων, χωρίς τροπολογίες. Πρώτη παράγραφος. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερη παράγραφος υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 5. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ε. Αιτιολογική σκέψη του προημίου. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Το σύνολο του κοινοψηφίσματος. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. ψηφοφορία τεσσάρων προτάσεων ψηφίσματο με θέμα τον εξοχρονισμό τη νομοθεσία στον τομέα του ΦΠΑ, ώστε να δοθεί όθηση στην ενιαία ψηφιακή αγορά. Κοινό σχέδιο ψηφίσματο τριών πολιτικών ομάδων, χωρί τροπολογίε. Ψηφίζουμε το σύνολο του ψηφίσματο με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλο ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Επόμενη έκθεση, έκθεση του κυρίου Λίσεκ με θέμα της διαπραγματεύσεις για τη Συμφωνία Σύνθεσης, Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Γεωργίας. Σχέδιο ψηφίσματος. Τροπολογία 7. Ποιος είναι υπέρ. Διαδικαστικό, συγγνώμη, ο εισηγητής ο κύριος Ξιστόφ Λίσεκ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Μια στιγμούλα μόνο θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ βάθους καρδίας όλους τους και ηγητές, αλλά και τα θεσμικά όργανα που συνέβαλαν στην εκπόνηση τη έκθεση αυτή. Θα ήθελα να σα πω ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η έκθεση, όχι μόνο για μας, για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά πρόκειται για έκθεση που περιμένουν διακαώς και η κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο και σύσσωμο ο λαός της Γεωργία. Σας ευχαριστώ τραπολογία 7. είναι υπέρ? κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3 ποιος είναι υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 4. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 6. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Ο κύριος Βομπότα θα υποβάλει προφορική τροπολογία στην τροπολογία 5. Παρακαλώ κύριε Βομπότα, έχετε το λόγο Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω υποβάλει μια τροπολογία εξ ονόματος της ομάδας μας θα, η οποία ήταν ε, κάπως ακατανόητη. Θέλω να αντικατασταθεί από την εξή και ελπίζω να συμφωνήσουν οι συνάδελφοι καλεί τις αρχές της Γεωργίας να μην χρησιμοποιούν ανάλογη πολιτική πίεση εναντίον των πολιτικών αντιπάλων της κυβέρνησης. Υπενθυμίζει πως ένα ανταγωνιστικό και αποτελεσματικό πολυκομματικό σύστημα είναι ουσιαστικό για την εδραίωση της δημοκρατίας στη Γεωργία. Ευχαριστώ. Μάλιστα υπάρχουν ενστάσεις για την προφορική τροπολογία. Φαίνεται ότι ε, είναι αρκετή. Δυστυχώς, κύριε Σβόμποντα, δεν μπορούμε να ψηφίσουμε την προφορική τροπολογία. Καλώς. Ελπίζω να μην υπάρχει πρόβλημα με την ουσία της ε, τροπολογίας, την πολυκομματική δημοκρατία δηλαδή θα ήθελα να αποσύρω και την αρχική μου τροπολογία γιατί η έκθεση του συναδέλφου είναι πάρα πολύ καλή έκθεση και δεν θα πρέπει να περιέχει στοιχεία που δίνουν λάθος πληροφορίες. Οπότε αποσύρω την αρχική τροπολογία για να μην χρειαστεί να την ψηφίσουμε. Ευχαριστώ. Ε, so, Αν κατάλαβα καλά, αποσύρετε την τροπολογία 5. Ε, εντάξει, δεν θα ψηφίσουμε Ψηφίζουμε το σύνολο του σχεδίου ψηφίσματος με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Επόμενο θέμα. Ε, συγχαρητήρια κύριε Λίσεκ και σας ευχαριστούμε. Να μην το ξεχάσω. Επόμενο θέμα, έκθεση Γκούσταυσον με θέμα την εσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σχέδιο ψηφίσματος χωρίς τροπολογίες. Παράγραφος 2, σημείο ε. Τα κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα, ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, ποιος είναι υπέρ. Κατά Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για το δεύτερο τμήμα της παραγράφου 2 σημείο ε. Άρχεται η ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Εγκρίνεται το πρώτο τμήμα. Ε, παράγραφος 2 από σημείο G. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 4. Ψηφοφορία κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για το δεύτερο τμήμα της τέταρτης παραγράφου. Με ηλεκτρονικό έλεγχο. Παρακαλώ, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 6. Ψηφοφορία κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. ποιο είναι υπέρ στο δεύτερο, για το δεύτερο τμήμα. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 11. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 12. Κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την παράγραφο 12, το πρώτο τμήμα συγκεκριμένα, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλο. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται και αυτό. Ηλεκτρονικός έλεγχος για το δεύτερο τμήμα της παραγράφου 12. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Από το προήμιο, το νη. Ποιος είναι υπέρ. Αιτιολογική σκέψη νη. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται και το σύνολο του σχεδίου ψηφίσματος με ονομαστική κλίση άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ευχαριστούμε τον κύριο Γκούσταυσο. Επόμενο θέμα, έκθεση της κυρίας Λεύιν με θέμα την καταπολέμηση της παράνομης αλίας στο παγκόσμιο, σε παγκόσμιο επίπεδο και το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σχέδιο απόφασης χωρίς τροπολογίες. Ψηφίζουμε. Παράγραφος 12, πρώτο τμήμα. Άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται δεύτερο τμήμα, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 13. Πρώτο τμήμα, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Άρχεται ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία. Επαναλαμβάνω. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 33. Άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Η κυρία Λεύιν έχει μια προφορική τροπολογία για την παράγραφο 35. Έχετε το λόγο, κυρία Λεύιν. Ευχαριστώ πολύ. Θα θέλαμε να αφαιρέσουμε τη λέξη στην ε, αρχή της παραγράφου 35 και να την αντικαταστήσουμε με τις λέξεις examine the possibility of adding, να εξετάσει την, ε, το ενδεχόμενο της προσθήκης και να συνεχίσουμε λαμβάνοντα τα μέτρα για την ε, ε, διατήρηση των ελευθερικών αποθεμάτων ε, σύμφωνα με τις διαδικασίες και το κάνουμε αυτό γιατί δεν θέλουμε να προδικάσουμε οποιαδήποτε απόφαση της αρμόδιας επιτροπής και ελπίζω ότι θα δεχτείτε αυτή την προφορική τροπολογία. Σας ευχαριστώ. Υπάρχουν αντιρρήσεις για την προφορική τροπολογία? Όχι. Ψηφίζουμε την παράγραφο 35 με την προφορική τροπολογία. Ποιο είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφο 40. Ποιο είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Το σύνολο του ψηφίσματος άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται σας ευχαριστούμε και συγχαρητήρια κυρία Λέβιν. Ολοκληρώσαμε τις ψηφοφορίες. Σας ευχαριστώ και ραντεβού σε δύο εβδομάδες ε, στην Ολομέλεια.